Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι στην απογευματινή μας αυτή συνεδρίαση. Ε, είναι ασύνηθες να συνεδριάζουμε πέμπτη απόγευμα. Η Επιτροπή Γεωργίας τουλάχιστον πολύ σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, αυτή είναι μία από τις σπάνιες φορές και μάλιστα έτυχε και να είναι σε περίοδο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές. Εξού και η σχετικά χαμηλή παρουσία, μικρή προσέλευση των Ευρωβουλευτών. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα την πεμπτουσία τουλάχιστον των όσων θα ακούσουμε σήμερα θα τα μεταφέρουμε και στους συναδέλφους. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης χωρίς παρατηρήσεις εγκρίνεται. Σημείο 2. Έχουμε μετάδοση απευθείας στο διαδίκτυο και έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. Οπότε περνάμε στο κυρίως θέμα, το σημείο 3, τη δημόσια ακρόση με θέμα την ε, γενετική ποικιλότητα, ποικιλομορφία, την διατήρηση και των ε, καλλιεργειών με τους συγγενείς ε, οργανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της βιοπικιλότητας και γι' αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους εμπειρογνώμονες που αποδέχθηκαν ε, την πρόσκληση της Επιτροπής και ήρθαν να μας διαφωτίσουν. Ε, ξέρετε ότι έχουμε την στρατηγική για την βιοπικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2001 που προσδιορίσε φιλόδοξους στόχους και δράσεις για να αναχαιτιστεί η απώλεια βιοπικιλότητας ε, στη Γεωργία και η απώλεια των ε, υπηρεσιών οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή αυτή θα συμβάλλει στο να ε, αναχαιτιστεί η απώλεια και της παγκόσμιες βιοπικιλότητας μέχρι το 2020. Έχουμε μια σειρά υποχρεώσεων που μας δεσμεύουν, όπως και την σύμβαση του 2010, τη Διεθνή Σύμβαση για την Βιολογική Ποικιλότητα. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα στις αρχές του 2016 ε, με στόχο να επικεντρωθούμε στις ε, υψηλές προτεραιότητες προκειμένου να ε, υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα άγρια συγγενή των καλλιεργούμενων φυτών, τη την διαφύλαξη των τραπεζών γονιδίων, το ρόλο της γενετικής βιοπικιλότητας, Ω προ την επιστηστική ασφάλεια και τη βιοποικιλότητα, γιατί πραγματικά τα άγρια συγγενή καλλιεργούμενων φυτών ε, ε, είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι, ε, έχουν ε, πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα καλλιεργούμενα φυτά, αλλά ε, βλασταίνουν με φυσικό τρόπο σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Γι' αυτό μπορούμε να τα διασταυρώσουμε με υπάρχουσες καλλιέργειες για να είναι πιο ανθεκτικές και να προσαρμόζονται καλύτερα στις τοπικές συνθήκες και να είναι και πιο ανθεκτικές κλιματικές αλλαγές. Μας ενδιαφέρει αυτό, να διατηρήσουμε δηλαδή, να διαφυλάξουμε τέτοια είδη σε ασφαλείς τράπεζες γονιδίων αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και τα φυσικά ενδιατήματά τους, ώστε να συνεχίσουν να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή δημόσια κρόση θα μας επιτρέψει να εγγύψουμε πιο σχολαστικά σε αυτά τα θέματα και να δούμε πώς ε, θα τροποποιήσουμε και μετά το 2020 προς αυτή την κατεύθυνση και την κοινή γεωρική μας πολιτική. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους καλεσμένους μας. Τη σειρά την έχουμε ήδη κανονίσει. Πρώτα θα λάβει το λόγο ο καθηγητής Νάιτζελ Μάξτετ από, το, από τη Σχολή Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιχαμ, που είναι ο κύριος Μάξτε είναι λέκτορ σε θέματα γενετικής διατήρησης με ιδιαίτερες γνώσεις για τις τεχνικές διατήρησης in situ και ex situ και επίσης συμμετέχει στη γνωμοδοτική ομάδα για την παγκόσμια γεωργική έρευνα. Καλώς ορίσατε. Δεύτερη ομιλήτριά μας είναι η κυρία Σούζαν Μπέρθ, δόκτωρ Σούζαν Μπέρθ, από το Εθνικό Ελλαδικό Πρόγραμμα για την Έρευνα στις Καλλιέργειες. Καλώς ήρθατε. Ασχολείται με είδη χορτονομής, ε, ε, ζυζάνια και δημητριακά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους γενετικούς πόρους και τις ε, δραστηριότητες γονιδιωματικής. Μάλιστα από το 2009 είναι και εκδότρια η δόκτωρ Σουζαν Μπέρθ του περιοδικού «Τα χρονικά της βοτανικής». Καλώ ήρθατε κι εσεί. Και τρίτος μα ομιλητής θα είναι ο δόκτωρ Νίκολα Γου, ε, επιστήμονα Ερευνητή ε, και συντονιστή ε, του Bioversity International στο Μομπέλιε τη Γαλλία, Επικεντρώνεται σε θέματα γενετικών πόρων και γονιδιωματικής φυτικών διαδεδομένων καλλιεργιών, συμπεριλαμβανομένων και των πανανών από το 2011. Μάλιστα είναι συντονιστής του Παγκόσμιου Δικτύου Διατήρησης των Γενετικών Πόρων της Μπανανιάς και του Μούσανετ του Δικτύου για την Μπανανιά. Και επίση ενεργό μέλο τη της ομάδα Ομάδας Διεθνούς Δικτύου Γεωργικής Έρευνας. Έχετε γύρω στα 10 με 15 λεπτά το πολύ όμω για τις παρεμβάσει των εμπειρογνωμόνων. Παρακαλώ θερμά να μην υπερβείτε το τέταρτο και θα ακολουθήσει μετά από κάθε παρουσίαση συζήτηση με υποβολή ερωτήσεων από την Ομίγυρη. Θέλουμε στις 4 να ολοκληρώσουμε τη δημόσια κρόση, οπότε χρόνο έχουμε. Διερμηνή έχουμε μέχρι τις 4, γι' αυτό μέχρι τότε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Χαιρετίζω από ευκαιρία και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Και περνάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για την σημασία των άγριων συγγενικών καλλιεργιών και πώς το ζήτημα αυτό σχετίζεται με τις στρατηγικές διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό και οι σχετικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχά θα πρέπει να σα πω ότι έχουμε έναν ανθρώπινο πληθυσμό ο αυξάνεται συνεχώ. 7,5 δισεκατομμύρια είναι τώρα το 2017 και 78% ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα φτάσουμε τα 9,8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Το 86% των οποίων, των ανθρώπων αυτών, θα ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί βέβαια χρειάζονται τρόφιμα. Για να θρέψουμε λοιπόν τον παγκόσμιο πληθυσμό μέχρι το 2050, χρειάζεται να αυξηθούν κατά 60% ε, ο εφοδιασμός σε τρόφιμα, ενώ 100% θα πρέπει να αυξηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέχρι το 2050 όμως θα μειωθεί και η γεωργική παραγωγή εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, μάλιστα με ένα ρυθμό 2% κάθε δεκαετία. Θα έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά μία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και από την άλλη μία μείωση τη γεωργική παραγωγή εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Τα αριθμητικά δεδομένα που βλέπετε στο κάτω μέρο τη διαφάνεια αντιστοιχούν ουσιαστικά στα αριθμητικά αυτά δεδομένα. Μία πρόσφατη έρευνα που έκανα στο ΜΑΝ καταδεικνύει αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει με το Made Gatus Katavi, το οποίο είναι ένα άγριο συγγενικό είδος με κόκκινο μπορείτε να δείτε τώρα πού μπορεί να καλλιεργηθεί το ΑΑ, 12% του ΟΜΑΝ. Μέχρι το 2020 όμως προβλέπεται ότι η περιοχή αυτή θα αυξηθεί. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν βλέπουμε μια αύξηση στην παραγωγή ΑΑ. Αυτό για το 2020. Δείτε όμως πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το 2050. Η ε, επικράτεια όπου μπορεί να καλλιεργηθεί το είδος αυτό φτάνει το 2,3% μόνο. Αυτό ενδεχομένω να ακούγεται κάπως ακραίο, αλλά καταδεικνύει τελικά πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τα, παράτητα, τα απαραίτητα γονίδια προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλλιέργεια αυτού του είδου. Αν λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε την παραγωγή στο συγκεκριμένο αυτό είδος ή και σε άλλα είδη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις στρατηγικές βιοπικιλότητας που μας προσφέρουν τα είδη άγνωση συγγενικών καλλιεργειών. Πρόκειται ουσιαστικά για τους άγριους προγόνους κάποιων φυτών και το θετικό είναι ότι μπορούμε να μεταφέρουμε γονίδια από τα άγρια είδη προς τα καλλιεργήσιμα είδη. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ανθεκτικότητα των φυτών αυτών σε διάφορους επιβλαβείς οργανισμούς. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη βιοπικιλότητα εκτός του καλλιεργήσιμου είδους. Βλέπετε εδώ πέρα ένα άγριο συγγενικό είδος του σιταριού όπου στο αριστερότημα της διαφάνειας βλέπετε περίπου 50 διαφορετικά άγρια συγγενικά είδη του ΣΥΤΟΥ, ενώ στην κεντρική στήλη βλέπετε ένα κατάλογο από διάφορα χαρακτηριστικά που μπορείτε να έχετε από αυτά τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Και αν μεταφέρετε το συγκεκριμένο γονίδιο από το άγριο συγγενικό φυτικό είδος προς το καλλιεργήσιμο σύτο... καταφέρνει να πετύχεται μία ανθεκτικότητα του φυτού και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε επίσης και την παραγωγή και τη σοδιά. Καθότι Μιλάω τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένω ενδιαφέρει και η χρηματοοικονομική πτυχή του ζητήματο. Όσον αφορά την ετήσια αξία τη μεταφορά των γονιδιακών χαρακτηριστικών από το άγριο είδος προς το καλλιεργήσιμο είδος, το 1997 έγινε μια εκτίμηση ότι, όπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως θα μπορούσαν να προκύψουν στα πλαίσια της αύξησης της ε, καλλιεργήσιμης παραγωγής, αν χρησιμοποιηθούν τα γονίδια αυτά. Πιο πρόσφατα, το 2013, η PricewaterhouseCoopers έκανε μία ανάλογη μελέτη, αλλά αυτή την φορά για, για τα 29 μεγαλύτερα καλλιεργήσιμα είδη και πάλι κατέληξε σε αυτό το ποσό, σε αυτή την αποτίμηση, 150 δισεκατομμύρια. 115 με συγχωρείτε δισεκατομμύρια. Μολονότι το ποσό αυτό φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν δείτε τη γραφική παράσταση στο δεξί τμήμα της διαφάνειας, βλέπετε εδώ πέρα ότι μιλάμε για διαφορετικές καλλιέργειες και η στήλη που βλέπετε εδώ πέρα έχει να κάνει με το διαφορετικό είδος τελικά. Βλέπετε ότι αν για παράδειγμα βγάλετε εκτός τα πρώτα 10 φυτά, υπάρχει μια περιορισμένη τελικά, πολύ περιορισμένη χρήση των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών στις καλλιέργειες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι η συνολική αξία αν χρησιμοποιηθούν τα άγρια συγγενικά φυτενικά είδη, θα είναι 300 δυνάμει, 300 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αν τελικά χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα άγρια συγγενικά είδη και αν επεκτείνουμε τη χρήση τους και σε άλλα είδη, όχι μόνο σε αυτά τα οποία εμφανίζονται σε αυτή τη γραφική παράσταση. Προφανώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια αυτά αν δεν είναι διαθέσιμα. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν καταρχάς είναι τι συμβαίνει με τις απειλές και τι συμβαίνει με το ζήτημα της διατήρησης. Μία μελέτη που έγινε από το IUCN πριν από μερικά χρόνια έδειξε ότι ένα 16% των ειδών αυτών στην Ευρώπη εξέτασε περίπου 572 τέτοια άγρια γενικά φυτικά είδη και είπε το 16% απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ ένα 4% κινδυνεύει με εξαφάνιση. Αυτά όσον αφορά την πτυχή της απειλή, Όσον αφορά τώρα την πτυχή της διατήρησης. Όσον αφορά την εκτόπου διατήρηση, την εξή, του διατήρηση, έχουμε δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι συγκεκριμένα για την Ευρώπη. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες βάσεις, κάποιες τράπεζες γονιδίων και περίπου το 1 τρίτο δεν εκπροσωπείται καθόλου σε αυτές τις τράπεζες γονιδίων. Περίπου ένα τρίτο πάλι, για ένα τρίτο υπάρχει, υπάρχουν μόνο 10 καταχωρήσεις. Και πραγματικά θέλουμε να έχουμε μια πραγματική χρήση των γονιδίων των άγρων αυτών συγγενικών φυτικών ειδών, χρειάζονται 50 καταχωρήσεις, 50 εισαγωγές ανά είδος. Ένα τρίτο λοιπόν έχει μόνο 10 τέτοιες καταχωρήσεις και 72% ένα 72% των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών απαιτούν περαιτέρω συλλογή τέτοιων ε, ειδών, τέτοιων γονιδίων. Εξετάσαμε επίση και την επιτόπη διατήρηση, την in situ διατήρηση και είδαμε πάλι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελάχιστα τα μέρη εκείνα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια αποτελεσματική επιτόπια διατήρηση των άγρων αυτών συγγενικών φυτικών ειδών. Και μόνο σε μία περίπτωση για το ζαχαρότευτλο. Έχουμε και στην Ευρώπη, ε, στην Μαδέιρα, μια τέτοια τράπεζα γονιδίων. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πολύ περιορισμένη έξι του και in situ διατήρηση. Α δούμε τώρα ποια είναι η πολιτική η οποία ακολουθείται, ποιο είναι το πλαίσιο πολιτική. Είναι αρκετά παγιωμένο, θα έλεγα. Γίνεται μια αναφορά στο στρατηγικό σχέδιο τη CBD, όπου γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη διατήρηση των άγρων συγγενικών καλλιεργιών λέγεται συγκεκριμένα ότι στον στόχο 9 ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη και αυτό συνδέεται άμεσα επίσης και με τους στόχους της χιλιετίας, κυρίως στον στόχο 1, 2, 3, συγγνώμη, το διαβάζω πολύ καλά, προκειμένου να καταφέρουμε να εξελίψουμε τη φτώχεια, να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη επιστηστική ασφάλεια, καθώς επίσης και την ευημερία των πολιτών. Βλέπετε λοιπόν ότι τα άγρια συγγενικά φυτικά ήδη συνδέονται επίση και με την επίτευξη αυτών των στόχων. Σα είπα ότι δεν έχουμε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά την Ευρώπη, αλλά πρόσφατα σε παγκόσμιο επίπεδο η νορβηγική κυβέρνηση έκανε μία μελέτη. Ξέρετε ότι η νορβηγική κυβέρνηση έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ στο Global Crop Diversity Trust προκειμένου να προωθήσει περισσότερο την μη επιτόπια συλλογή τέτοιων άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Εγώ με την ερευνητική μου ομάδα προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε τα πιο σημαντικά αυτά άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Στη συνέχεια κάναμε μια ταξινόμηση των δεδομένων αυτών και προσπαθήσαμε να δούμε πού βρίσκονται τα ίδια αυτά και από πού θα μπορούσαμε να τα συλλέξουμε. Όσον αφορά λοιπόν πιο συγκεκριμένα την Ευρώπη, Βλέπετε 31 χώρες στην Ευρώπη που έχουν πάνω από 20 από τα άγρια αυτά συγγενικά φυτικά είδη που αποτελούν προτεραιότητα. Οι πρώτες χώρες είναι η Ιταλία, η Ισπανία και ακολουθούν και κάποιες άλλες χώρες όπως βλέπετε. Όσον αφορά τώρα το παγκόσμιο τέτοιο αριθμό άγριων συγγενικών καλλιεργιών, έχουμε 1392 τέτοια είδη προτεραιότητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μα εδώ πέρα στην Ευρώπη. Βλέπετε εδώ πέρα τον επιμερισμό, την κατανομή αυτών των ταξινομικών ομάδων για τα άγρα συγγενικά φυτικά είδη. Βλέπετε επίση που υπάρχει μία επικάλυψη. Βλέπετε ξεκάθαρο ότι όσον αφορά την Ευρώπη, ότι οι πορτοκαλί και οι κόκκινε περιοχέ εμφανίζονται κυρίω στη Μεσόγειο, στην ακτή τη Μεσογείου σε διεθνέ λοιπόν παγκόσμιο επίπεδο, οι περιοχέ όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων άγρων συγγενικών φυτικών ειδών και όπου υπάρχει ε, ουσιαστικά μια πολύ σημαντική οικονομική αποτίμηση, αν θέλετε, των ειδών αυτών, είναι η περιοχή τη ε, Μεσογείου. Εδώ πέρα βλέπετε πού προκύπτουν κάποια κενά όσον αφορά τη διατήρηση, πού δεν έχουμε κάνει επαρκή συλλογή τέτοιων ε, ειδών. Και πάλι βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες ευκαιρίες στην Ευρώπη και ιδίως στις μεσογειακές χώρες ή ακόμα και στην Νότιο Αμερική. Στο... Στην Νότια Αμερική βλέπετε εδώ πέρα συγκεκριμένε αιστείες συλλογής των φυτών αυτών, καθώς επίσης και στην Ινδονησία. Και εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε πολλά άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε που μπορούμε να κάνουμε in situ διατήρηση. Σε κάθε μία από τις βούλες που βλέπετε στο χάρτη αυτόν έχουμε τόπους όπου θα μπορούσαμε κατά προτεραιότητα να έχουμε in situ διατήρηση για τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Και βλέπετε πάλι εδώ στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Μεσόγειο περίπου το ίμιση των ε, εστιών αυτών εντοπίζεται, των παγκόσμιων αυτών εστιών εντοπίζεται στην περιοχή της Ευρώπης και της ε, Μεσογείου, καθώς επίσης και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε στην Ευρώπη να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο με την ε, διατήρηση αυτήν. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης και της συλλογής και ιδίω όσον αφορά το πρόγραμμα για τη διατήρηση των γενετικών πόρων και της γενετικής ποικιλομορφία, το οποίο επικεντρώνεται και σε άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Θεωρώ ότι ο οργανισμός αυτός από τότε που συστήθηκε το 2000 έχει καταφέρει να αυξήσει πάρα πολύ την επαγγελματική και τη δημόσια ευαισθητοποίηση και μάλιστα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει και κοινοτική χρηματοδότηση. Τέσσερα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά συμβάλλουν πάρα πολύ στο να δημοσιεύονται διάφορες μεθοδολογίες και στο να φέρουν μαζί διάφορους ερευνητές από διάφορους χώρες πρόσφατα δημιούργησαν μία νέα στρατηγική, μία νέα νεολογική προσέγγιση όσον αφορά την διατήρηση των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Δεν θα ήθελα να σε εξηγήσω τώρα το διάγραμμα αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Καταδεικνύει πάντω ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι ότι η διατήρηση θα πρέπει να επιτελείται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν αιστείε όπου θα πρέπει να έχουμε κέντρα διατήρηση, αλλά θα πρέπει ανάλογε δομέ να έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται βέβαια από κάποιε πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η διατήρηση να οδηγεί και σε χρήση. Δεν υπάρχει λόγος να διατηρούμε τα πολύτιμα αυτά σπάνια άγρια συγγενικά φυτικά είδη αν στη συνέχεια δεν τα χρησιμοποιούμε. Ένα από τα τελευταία προγράμματα που προωθήσαμε στα πλαίσια του ECPC είναι το Farmer's Pride. Ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγκώνα στην Ιταλία μια πρώτη επαφή και ανταλλαγή απόψεων. Ουσιαστικά προσπαθούμε να γεφυρώσουμε εδώ πέρα διαφορετικέ κοινότητε. Καλλιεργητέ, βελτιωτέ φυτών, υπεύθυνου για τη διατήρηση των φυτών, μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το βασικό όμω πόρισμα τη συνεργασία αυτή θα είναι να πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την διατήρηση των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο και περισσότερο την κοινή γνώμη για τα ζητήματα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό συγκεκριμένο πλαίσιο στην Ευρώπη για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να το διερευνήσουμε το ζήτημα αυτό λίγο περισσότερο σήμερα. Όσον αφορά τώρα τις απαιτούμενε δράσεις, θα ήθελα τώρα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας πω εγώ τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε καλύτερη διατήρηση και χρήση των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Νομίζω ότι καταρχάς θα πρέπει να γεφυρώσουμε τα κενά τα οποία έχουν προκύψει. Να αναφερθώ καταρχάς στο κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή. Εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, πληρώνουμε προκειμένου να κάνω διάφορες δημοσιεύσεις, θα μπορούσα λοιπόν να υποβάλω πάρα πολλά έγγραφα στα οποία θα σας έλεγα πού και πώς θα πρέπει να γίνουν στρατηγικές διατήρησει. Αλλά στην πράξη όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία αν οι δικές μου θεωρητικές προσεγγίσεις δεν συνοδεύονται από μια έμπρακτη εφαρμογή των όσων προτείνω. Αναφέρθηκα πριν από λίγο σε ένα project το οποίο προωθήσαμε, το οποίο οδήγησε σε έναν κατάλογο γεωγραφικών χώρων όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τα κέντρα αυτά διατήρησης και δυστυχώς όμως αυτό δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο με την ισή του διατήρηση αν ακολουθούσαμε τα πορίσματα της έρευνας αυτής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην in situ και ex situ διατήρηση. Ένα 99% της χρηματοδότησης πηγαίνει στην ex situ διατήρηση. Το 99% της περιορισμένης χρηματοδότησης πηγαίνει στην ex του διατήρηση. 1% ενδεχομένω μόνο να προβλέπεται στην περιοχή της Μαδέιρα για την in situ διατήρηση. Αυτό προφανώς θα πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε επίσης να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στη βιοπικιλότητα και την αγροβιοπικιλότητα. Για ποιο λόγο το δίκτυο Natura 2000 να μην εμπλουτιστεί περισσότερο με πολιτικές και στρατηγικές που να έχουν να κάνουν με τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια διασύνθεση ανάμεσα στο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη διατήρηση των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή βιοπικιλότητα, θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης διατήρησης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ενσωματωθούν το τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αν θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα της έρευνας, θα πρέπει η διατήρηση να συνδεθεί περισσότερο με την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, με τον εντοπισμό συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και θα πρέπει στη συνέχεια ο καλλιεργητής ή ο βελτιωτής των φυτών να μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τα οποία του δίνουμε. Και ελπίζω ότι όλα τα πορίσματα της έρευνάς μας ουσιαστικά θα αναβαθμίσουν περισσότερο την προσέγγιση των πολιτικών σε σχέση με τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Αυτό είναι ένα μέρος μόνο των προτάσεων που θα μπορούσα να κάνω στη φάση αυτή. Όσον αφορά το τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι σαν τι μπαμπούσκε, τι ρωσικέ κούκλε, όπου το ένα εξαρτάται από το άλλο και το ένα ενσωματώνεται στο άλλο. Διάρθρωση τώρα τη διακυβέρνηση. Νομίζω το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει απαραίτητη διακυβέρνηση στην Ευρώπη όσον αφορά την in του διατήρηση. Αν σκεφτούμε λίγο την βιοπικιλότητα, έχουμε τους, τις διάφορες περιοχές Natura 2000. Δεν λέω ότι θα πρέπει κάτι αντίστοιχο να γίνει και για τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Ο στόχος μας είναι κάπως διαφορετικός. Οι χώροι Natura 2000 συνήθως έχουν να κάνουν με την παρουσία την απουσία κάποιων ειδών. Εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη διατήρηση της γονιδιακής ποικιλομορφία. Πρέπει να μπορούμε λοιπόν να διαχειριζόμαστε πλέον συγκεκριμένου χώρου στην Ευρώπη προκειμένου να εξασφαλίζουμε ακριβώς αυτή την βιοπικιλότητα. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε λίγο και το σύστημα των ε, σημαντικών ε, χώρων ε, φυτικής ζωικής κληρονομιάς όπου επιτελούμε συγκεκριμένε στρατηγικέ διατήρηση, ακριβώ επειδή τα ίδια αυτά είναι πολύ σημαντικά για τον επισητισμό. Τώρα το ECPGR, η επικεφαλής θεωρώ ότι βρίσκεται στην αίθουσα αυτή και ελπίζω ότι με ακούει. Οργανισμό αυτό έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική εργασία, αλλά δυστυχώ εξαρτάται μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των υπερογνωμόνων. Θα πρέπει να υπάρχει ο παρέτος μηχανισμό χρηματοδότηση προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να χρηματοδοτούμε την ε, Ευρωπαϊκή Διατήρηση Γονιδιακών Πόρων. Αυτή τη στιγμή ο οργανισμό αυτό έχει πολύ περιορισμένη χρηματοδότηση και δεν έχει την απαραίτητη πρόσβαση στην in situ και ex situ διατήρηση. Πρέπει επίσης να έχουμε μια γενικότερη, ένα γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο υποστήριξης. Και θα πρέπει να δούμε και λίγο τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους γονιδιακούς σπόρους για την μελλοντική παραγωγή τροφίμων και να υπάρξει ενδεχομένω και μια οδηγία για το ζήτημα αυτό. Περνάω και στη τελευταία μου διαφάνεια να σας πω λίγο μια δική μου προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν φοιτητή σε επίπεδο διδακτορικού, Βρισκόμουν στην νότια ακτή της Τουρκίας, ε, συνέλεγα εκεί πέρα διάφορα είδη και βρήκα ε, ένα νέο είδος ε, Το βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα αυτή. Ουσιαστικά σχετίζεται πάρα πολύ με το μπιζέλι. Ξέρετε ότι το μόνο χρώμα το οποίο μπορούμε να έχουμε στο άνθος είναι κίτρινο. Το ενδιαφέρον όμως στις νότιες ακτές της Τουρκίας είναι ότι το άγριο αυτό συγγενικό φυτικό είδος ε, είχε εν μέρη κίτρινα ε, λουλουδάκια. Επομένω θα μπορούσε όντω να χρησιμοποιηθεί, να διασταυρωθεί δηλαδή με το μπιζέλι. Εντόπισα το 1997 τον πληθυσμό του είδους αυτού, έκανα μια δημοσίευση και το 2005 τον επέστρεψα στην περιοχή αυτή της Τουρκίας, συμμετείχα σε μια συνδιάσκεψη, όχι αναγκαστικά πάλι για να ξαναδώ το είδος αυτό, πάντως ταξίδεψα στην περιοχή αυτή και με τρόμο είδα ότι ε, ο επιτόπου εκεί πληθυσμός του είδους αυτού είχε ουσιαστικά καταστραφεί, ακριβώς επειδή είχαν γίνει έργα στην περιοχή αυτή για να δημιουργηθεί ένα νέο αστυνομικό τμήμα. Επομένως, είχε καταστραφεί συνολικά όλο το ειδος αυτο αυτό. Ενώ είχαμε περίπου 20-25.000 τέτοια είδη, είχαμε φτάσει στα 5.000 μόνο. Ένα γεννητιστή θα σα πει ότι αυτό είναι το απόλυτο ελάχιστο προκειμένου να διατηρηθεί ένα απειλούμενο είδο. Είχα καταφέρει σε μία τράπεζα γονιδίων να περισσώσω τα γεννητικά χαρακτηριστικά του είδους αυτού και έγραψα ένα ακόμα άρθρο λέγοντας ότι η κατάσταση να πέσει, ότι προφανώς θα πρέπει να περισωθεί το είδος αυτό. Επέστρεψα πέρυσι για μια νέα συνδιάσκεψη και είδα το αστυνομικό αυτό τμήμα είχε επεκτηθεί και δίπλα στο αστυνομικό τμήμα χτίσανε και έναν επιπλέον δρόμο. Αυτή τη φορά λοιπόν κοιτώντα γύρω-γύρω την περιοχή, αντί για 25.000 ειδίδα, 15 μόνο. 15 τέτοια φυτά. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Βλέπετε εδώ πέρα ένα καταπληκτικό φυτό, το οποίο έχει μια τεράστια οικονομική αξία και εμεί εντελώ απερίσκεπτα το καταστρέφουμε. Αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε στο μέλλον τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Από τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διατήρηση. Γιατί δεν το ξεκινήσουμε αυτό τώρα, δεν πρόκειται να περισσώσουμε με τίποτα τα φυτά αυτά στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί συνδέεται άμεσα με την επισητιστική ασφάλεια. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντω πολύ πιστικά αυτά που μας είπατε. βέβαια, ε, μακρηγορήσατε κάπως, ξεπεράσατε το τέταρτο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Περάμε στη δεύτερη. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ε, να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου για το θέμα που μας απασχολεί. Θα σας πω πώ πώς τα βλέπει αυτά η Ιρλανδία από την ελλαδική σκοπιά που είναι ένα νησί στον Ατλαντικό και έχει ιδιαιτερότητες. Είναι και μικρή χώρα, αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο πλαίσιο και άλλων ε, μικρών ε, κρατών. Τα άγρια συγγενικά φυτά προς τα ημέρα ε, που καλλιεργούνται είναι πολύ συγγενή τα περισσότερα Ήμερα φυτά έχουν γονίδια και από τα άγρια. Στην Ιρλανδία χρησιμοποιούνται ε, τέτοια φυτά για να διασταυρώνονται και να δημιουργούνται νέα στελέχη πατάτας, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντική πηγή για να ε, διατηρηθούν βιώσιμα τα βιοσυστήματα για το μέλλον. Ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο ΦΑΟ, το 1995 είχε αναγνωρίσει σε μία έκθεση ότι στην ε, Ιρλανδία υπάρχουν ε, αυτόχθονα φυτά με γενοτύπους ε, που διατηρούνται λόγω της δυτικής θέσης και απομονωμένης. Αλλά δεν γνωρίζουμε ε, πάρα πολλά πράγματα για ε, τους γενετικούς ε, πόρους που υπάρχουν στα άγρια συγγενικά φυτά. Αυτό το πρόβλημα είναι κοινό και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και θαλάσσης είναι αρμόδιο για το συντονισμό και προώθηση μέτρων για τη διαφύλαξη και χρήση γενετικών πόρων για την γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. Υποστηρίζεται από μια Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Γενετικούς Πόρους όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες ενδιαφερομένων ΜΚΟ, πανεπιστημιακοί και Επίσης, εργαζόμενοι στο Υπουργείο συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Στην Ιρλανδία έχουν σημειωθεί 181 ε, συγγενικά, άγρια συγγενικά φυτά, 102 εκ των οποίων είναι ήδη που συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα 1 ε, δηλαδή τα φυτά αυτά που θεωρούνται προτεραιότητα για τη διαφύλαξη. Η διατήρηση εξ situ έχει αρχίσει και το Υπουργείο ε, Γεωργίας έχει τράπεζα σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, ιδιαίτερα για φύτα ενδυμικά και υπάρχει και ένα κέντρο για τη μελέτη της ε, πατάτας. Ε, πάνω από 400 ποικιλίε γεωμήλων έχουν ε, που συντηρούν και διατηρούν και in vitro και in situ. Στο Τσάκας εμείς έχουμε κάποια είδη που μελετούμε και διατηρούμε γιατί είναι πολύ σημαντικά για τη χορτονομή, για μια χώρα που εξαρτάται από τη βόσκηση στο ε, Trinity College του Δουβλίνου ε, υπάρχει τράπεζα γονιδιακή για απειλούμενα με εξαφάνιση φυτικά είδη της Ιρλανδίας. Ε, υπάρχει και ένωση στην Κομιτεία Κλέαρ και αλλού ενώσεις που ασχολούνται με τη διαφύλαξη και της φυτικής κληρονομιάς της Ιρλανδίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα συγγενικά αυτά είδη των καλλιεργούμενων φυτών. Στο 2010 δημιουργήθηκε το Εθνικό ε, Κέντρο Βιοπικιλότητα στο Γότερφορντ. Έχει πρωτογενείς πηγές δεδομένων από 55 τέτοια φυτικά είδη άγρια. Υπάρχει ε, το ε, η Εθνική Βάση Δεδομένων, το Εθνικό Βοτανολόγιο και Εθνική Δρυμή ε, και ε, Άγρια Πανίδα καταγράφονται σε ξεχωριστή τράπεζα δεδομένων. Επίσης, έχουν συγκεντρωθεί και άλλα στοιχεία από το Κέντρο Δεδομένων για την Εθνική Βιοπικιλότητα, καθώς επίσης και από όλα τα άλλα είδη. Ας πούμε υπάρχει βοτανολογική εταιρεία των Βρετανικών νήσων. Βλέπετε ε, ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα κέντρα και πώς υπάρχει η κατανομή ε, του ε, άγριους σπαραγγιού για παράδειγμα και άλλων ειδών. Επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό θα πρέπει να ενημερώνεται και το κοινό για το πόσο πολύτιμα είναι τα άγρια είδη, ε, ε, τα συγγενικά με τα καλλιεργούμενα. Ο Πολ ε, Κέρτης και ο Τόμ Κέρτης, συγγνώμη, και ο Πολ Γουίλαν έχουν μια υποστήριξη ακριβώς για να ενημερώνουν το κοινό και να αυξηθεί η συνειδητοποίηση για τη διατήρηση. Ένα νέο βιβλίο θα εκδοθεί το 18 την Άνοιξη. Επίσης, έχουν γίνει πολλές δημοσίευσεις ιδιαίτερα για τις πατάτες το 2008 και ε, για τα ε, ε, παραδοσιακά είδη μιλιάς το 2014. Υπάρχει Ε, επίσης για την Ήρα ε, μια επιστημονική εργασία. Για την πολυετή Ήρα. Βλέπετε τα στοιχεία αυτά με κόκκινο και πράσινο. Δεν ξέρω καταλαβαίνετε ακριβώς τι αναφέρεται εδώ. Είναι δύο βασικές κατηγορίες γονιδίων που μελετάμε. Τα δύο τρίτα ε, έχουν ε, ομοιότητες ε, με τα γονίδια που υπάρχουν πάντα για την Ήρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, ποια είναι η πραγματική πρόκληση από την διατήρηση in situ, επιτόπου. Έχουν γίνει κάποιες απόπειρες και έχει γίνει πάντως μια καλή αρχή για τα μήλα προσπαθούν ε, οι ε, αγρότες και οι ενδιαφερόμενοι να διαφυλάξουν τις διάφορες ποικιλίε, να διατηρήσουν το ε, αστικό υλικό και οι πατάτες, τα διάφορα είδη και οι σπόροι διατηρούνται σε ένα παράρτημα του Υπουργείου Γεωργίας. Πάντως, σε πολλά άλλα είδη ε, ε, όπως είναι οι ζωοτροφές ας πούμε, δεν έχουμε ε, τέτοια φαινόμενα. Είναι επίσης πολύ περίπλοκη και η διαδικασία της επικονίασης και τα έντομα που κάνουν την επικονίαση μειώνονται στην Ευρώπη. Για να διατηρηθεί λοιπόν σε ανοιχτά επίπεδα χρειάζεται πρόσοχη. Ιδιαίτερα για τη χορτονομή και χρειάζονται πρωτοβουλίες μακράς πνοής, καθώς επίσης και εργαλεία και όπλα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχουν ήδη ορισμένα και είναι πολύ μεγάλη η απειλή που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οικότοποι και βιότοποι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ε, με το άγριο τέφτλο που ε, ενδημεί ε, στην Ιρλανδία η διάβρωση των ακτών ή άλλες δραστηριότητες για χρήση γης, για οικοδομές κλπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απειλή για αυτό το είδος του τέφλου που φυτρώνει σε παραθαλάσσιες περιοχές η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη χρηματοοικονομικής υποστήριξη στην ε, διαφύλαξη των γενετικών πόρων, όλα αυτά είναι προβλήματα. Ένα ε, παράδειγμα του τεύτλου αυτού του παραθαλάσσιου, του άγριου, Αυτή είναι μια μελέτη που σας δείχνω. Που έχει μελετηθεί η κατάσταση από το 30, το 30, το 60 και το 80. Και εδώ βλέπουμε πόσες ε, περιοχές υπάρχουν που έχουν καταγραφεί από το 2007, από το 2 μάλλον μέχρι το 2007 και παντού σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει αυτό το τέφλο που φυτρώνει άγριο ε, και παρά την ε, άνηση κατανομή σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Στην surprisingly äh, ε, στο, στη βορειοδυτική Ιρλανδία έχουμε ε, έχουμε διάβρωση των ακτών και ανθρώπινη δραστηριότητα. Ε, υπάρχουν όμως περιοχές που θα πρέπει να καταδειχτούν ε, ως ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και το παραθέλαση αυτό ε, τέύτλο θα μπορούσε να θεωρείται ειδικού ενδιαφέροντος ε, φυτό η ποικιλία. Θα πρέπει όλες οι αρμόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης να γνωρίζουν ε, τα προβλήματα και να ξέρουν ότι στην περιοχή τους υπάρχουν άγρια είδη συγγενικά προς τα καλλιεργούμενα. Προχωρώ για, στην διατήρηση in situ για διάφορα είδη που έχουν να κάνουν και με το τοπίο γενικότερα ε, και τη διατήρηση του τοπίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, χορτονομή και για κάποια άλλα είδη. Ε, χρειάζεται ειδική προσέγγιση για να δούμε ποια είναι τα ειδικά οικοσυστήματα, οι βιότοποι και αν χρειάζεται να καλλιεργηθεί και η γη με τρόπο παραδοσιακό για να διαφυλαχθούν τα ντόπια είδη. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, ε, οι σωστές εκείνες πολιτικές μετά από ε, συνεργασία στην Ευρώπη των ερευνητικών ιδρυμάτων. Έχω κυκλοφορήσει εγώ μια ιδέα τέτοια στην ομάδα εργασίας Τσάγκας για την βιοπικιλότητα Ε, όπως η εθνική δρυμή ας και η προστασία της άγριας πανίδας ε, και χλωρίδας. Οι αγρότες θα πρέπει να αμείβονται ε, για να διατηρούν αυτά τα φυτά και να μην τα εκριζώνουν. Άρα χρειάζεται ε, μια πρακτική μακράς πνοής ε, με στόχο τη διαφύλαξη αυτών των ειδών και τη διατήρησή τους. Ας πούμε, στην κοινή γεωργική πολιτική ενδεχομένως να ε, μπορούν να συμπεριληφθούν και τέτοια μέτρα. Αλλά αυτά έχουν συνήθως ορίζοντα πενταετίας ή επταετία στα προγράμματα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό δεν αρμόζει σε μια διαφύλαξη και διατήρηση ειδών χορτονομής. Στην Ελβετία και στην Νορβηγία, ωστόσο, έχουν επιτευχθεί προοδοί. Θα μας πείτε τώρα ότι είναι βέβαια οι πλουσιότερες χώρες στην Ευρώπη. Ναι, αλλά ε, έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα ωφέλη προς τους αγρότες, έχει δείξει ότι ε, τα ε, βοσκοτόπια, οι μικτές καλλιέργειες είναι πάρα πολύ πιο αποδοτικές με πολύ μεγάλη ε, απόδοση συγγνώμη, παρά να είναι μόνο καλλιέργειες. Αυτό συνηγορεί και υπέρ της ε, διατήρησης των άγριων συγγενικών ε, ειδών και μπορούν να ενταχθούν αυτά τα μέτρα στην κοινή γεωργική πολιτική ενδεχομένως. Uh, uh, uh, Το 1999 δημοσιεύθηκαν σχετικά αποτελέσματα. Συμπεράσματα και περίληψη. Υπάρχουν ε, διάφορες συλλογές, έξι του για τη διαφύλιση, αλλά σε πολύ ε, μικρούς αριθμούς, εξαιρετικά μικρούς αριθμούς για συγκεκριμένα είδη και ε, μάλλον αυτό μπορεί να μην είναι βιώσιμο στο δίνικες αν δεν υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός ε, ρηγμάτων. Η έξι του διατήρηση είναι πάρα πολύ ε, ακριβή, έχει ένταση εργασίας, χρειάζεται πολύ ποιοτικό έλεγχο και ε, ταξινόμηση του υλικού που αποθηκεύεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης όμως να το έχουμε. Δεν είναι ο μόνος τρόπος διατήρησής μας. Επίσης έχουμε στείλει στο Σφάρμπαρτ ε, υλικό για τη χορτονομή και τη βατάτα. Είναι εξαιρετικό αυτό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συλλογή. Χρειάζεται συνεχή ενημέρωση όμως το σύστημα ε, των σπόρων που διατηρούνται στο Σφάλμπαρτ. Είναι μια πρωτοβουλία των κρατών μελών, αλλά ε, μπορεί να προωθηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές στις διάφορες χώρες και οι φορολογούμενοι τι κάνουμε και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα ε, χρήματά τους. Υπάρχει και μια στρατηγική ή στρατηγικές για τη διατήρηση in situ επιτόπου. Αυτά έχουν μείνει πίσω. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να ε, διατηρήσουμε τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές για να διαφυλάσσουμε την ποικιλία των ειδών. Ωστόσο, ο έλεγχος των στρατηγικών αυτών ε, απαιτείται, ιδιαίτερα για τα απειλούμενα είδη και χρειάζεται να αναπτύξουμε μέτρα και πολιτικές ε, για την διατήρηση των συγκινικών αυτών ειδών επιτόπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα μικρό ταμείο που υπάρχει ε, στην ε, Ιρλανδία που έχει ένα προπολογισμό 50.000 ευρώ για τη διαφύριξη ε, αυτού του υλικού και δεν ασχολείται μόνο με φυτά αλλά και με είδη εντόμων και ζώων. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε και, και πιο μικρές ΜΚΟ όταν ζητούν χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές τους. ήθελα επίσης να ευχαριστήσω διαφόρους συναδέλφους από την Ιρλανδία που με βοήθησαν να συγκεντρώσω όλα αυτά τα στοιχεία για τη σημερινή παρουσία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάρθ. Και δίνω το λόγο στον τρίτο και τελευταίο καλεσμένο μας, τον κύριο Νικολάρου. Ε, χρόνου φίδου. Ναι, θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω καν το τέταρτο. Νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας ε, για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι η γενετική βιοπικιλότητα που είναι ζωτική σημασία για την ε, επιβίωση του ανθρώπινου γένους, του ανθρώπινου είδου των φυτών, της Χλωρίδα και τη Πανίδα. Και σα ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνετε να σα μιλήσω για την ε, διατήρηση και τη χρήση της αγροβιοπικιλότητας για καλύτερα τροφικά συστήματα. Μάλιστα θα ασχοληθώ με μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα, θα σας αναλύσω την περίπτωση της μπανάνας που δεν είναι ένα ε, προϊόν ε, της Ευρώπης παρόλο που έχουμε μικρή παραγωγή και στην Ελλάδα και την Ισπανία αλλά είναι το προϊόν που καταναλώνουμε κατά κόρον στην Ευρώπη παρόλα αυτά. Θα ήθελα καταρχήν να σας μιλήσω για την οργάνωση στην οποία δουλεύουμε. Είναι η Bioversity International που είναι ε, τμήμα ενός ομίλου από 15 ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο και τα κέντρα αυτά υπάρχουν εδώ και μία πεντηκονταετία από την πράσινη, την οικολογική δηλαδή επανάσταση που αναπτύχθηκε από τον Όρμαν Μπαλόν βραβευθέντα με βραβείο Νόμπελ. Είμαστε η μόνη οργάνωση που έχει παραρτήματα και γραφεία ανά τον κόσμο. Μάλιστα έχουμε γραφείο και στην Ευρώπη και όπως βλέπετε στη φωτογραφία τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Ρώμη αλλά έχουμε υποκατάστημα στο Μομπελιέ όπου διαβιώ εγώ και ένα τμήμα του γραφείου μας ε, βρίσκεται στη Λέβεν, λίγα χιλιόμετρα από εδώ δηλαδή και έχουμε εργαστήριο με τη μεγαλύτερη δεξαμενή γονιδίων μπανάνας Έχουμε όμως και κάποιους ε, επιστήμονες συνεργάτες μας στην Ισπανία. Σκοπός μας και η αποστολή μας είναι να δώσουμε επιστημονικές αποδείξεις ε, πρακτικές διαχείρισης και επιλογές πολιτικής για να χρησιμοποιούμε και να διαφυλάσσουμε την ε, γεωργική και βιοπικιλότητα της Πανίδας, που είναι πολύ σημαντική. Η αγροβιοπικιλότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπε και ο πρώτος εμπειρογνώμονας. Ε, και μάλιστα όχι η βιοπικιλότητα γενικά, ειδικά η αγροβιοπικιλότητα είναι πολυεπίπεδη. Σε επίπεδο κατανάλωσης ενδιαφέρει την ανθρώπινη υγεία, γιατί η ποικιλομορφία, η πολυμορφία του φαγητού είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική και για τι αγορέ, για καλύτερο βιοπορισμό, στην παραγωγή, για βιώσιμη γεωργία και υπηρεσίε οικοσυστήματος, αλλά και για του γενετικού πόρου, για την προσαρμογή και την ανανέωση εδώ στη μέση της γραφικής παράστασης έχουμε όλες αυτές τις συνιστώσεις που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, άρρηκτα συνδεδεμένες. Γι' αυτό μπορούμε να διαχειριστούμε και να προωθήσουμε την αγροβιοπικιλότητα ε, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο διατήρησης παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο αγοράς και κατανάλωσης. Και για να διαθήσουμε επιχειρήματα αυτά που σας είπα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την περίπτωση της μπανάνας και γιατί διαλέξαμε τις μπανάνες, γιατί είναι η 8η παγκοσμίω σημαντικότερη καλλιέργεια και όταν α, λέω μπανάνα δεν εννοώ αυτή της φωτογραφίας αλλά και τις μπανάνες μαγειρικής, plantains και όχι μόνο αυτές που τρώμε ως φρούτα και ένα μεγάλο τμήμα τους καλλιεργείται και στην Λατινική Αμερική. Πάντως ε, το μεγαλύτερο τμήμα της ε, παραγωγής είναι μπανάνες τύπου Cavendish, ενός είδους δηλαδή, και περίπου το 50% εξαρτούνται από ένα και μόνο κλόνο, ένα και μόνο στέλεχος. Ε, η διάβρωση της βιοπικιλότητας αυξάνεται καθημερινά και αυτό αυξάνει και την ευπάθεια σε επιβλαβείς οργανισμούς και ε, νόσους. Είχαμε την περίπτωση της, ε, του λοιμού λόγω της έλλειψης ε, πατάτας που αποδεκατίστηκε από ένα επιβλαβή οργανισμό. Πριν από μία 50 κονταετία είχαμε όξυση της, του επιπολασμού της φουζαρίωσης της νόσου του Παναμά που ήταν μία θανατηφόρος με που ρήμαξε πραγματικά τις εξαγωγές πρόκειται μια, για μια μικητίωση που περνάει μέσα από το έδαφος και πλήττει τα αγκία του φυτού. Και μάλιστα η ποικιλία Κάβεντις, που είναι πια η δεσπόζουσα ποικιλία, και μάλιστα κατά τύχη βρέθηκε στα, στη, νότια, Κίνα και στο Βιετνάμ στις δεκαετίες του 60 και 70 έχουν, έχει αντικαταστήσει την προηγούμενη ποικιλία που ήταν η κρατούσα και στις τοπικές και στις μπανάνες εξαγωγής και μάλιστα το νέο στέλεχος που ρέκεψε στη δεκαετία του 90 είναι η Tropical Race For και είχε αποδεκατήσει την Κάβεντι στην Ασία, Ειρηνικό και Αφρική και μάλιστα μόλις επέστρεψα από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική από ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 300 παραγωγοί και ερευνητές και εκεί συζητήσαμε πώς θα αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα πώς θα αποτρέψουμε τη μετάδοση της νόσου αυτής από τη μία ήπειρο στην άλλη. Ε, υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες. Ε, με 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε την επέλαση αυτής της Ρώσου και να δούμε ποια είναι τα ανθεκτικά στελέχη. Αν δεν κάνουμε όμως τίποτα θα μας στοιχήσει 10 δισεκατομμύρια. Ενώ εκατομμύρια θα ήταν το κόστος του να βρούμε ανθεκτικό στέλεχος. Ε, οι ευρωπαϊκές αγορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο ρόλο στην αλλαγή αυτή τη κατάσταση. Μπορεί να σα εκπλήσει, αλλά το Βέλγιο είναι σημαντικότερο εισαγωγέ και επανεξαγωγέ μπανανών στην Ευρώπη. Περίπου ένα δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια διακινούνται από 40 περίπου εταιρείε. Βλέπετε εδώ τι πέντε σημαντικότερε χώρε εξαγωγή τη μπανάνα με βάση το τζίρο και τέταρτο παγκοσμίω είναι το Βέλγιο χάρη στη σημαντική θέση που έχει το λιμάνι της Αμβέρσας και τις σημαντικές εγκαταστάσεις και φυσικά μετά το Βέλγιο γίνεται ανακατανομή των φορτίων μπανάνας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόσφατα μάλλον διαπιστώσαμε με ενδιαφέρον σε μια τηλεοπτική εκπομπή ένα ντοκιμαντέρ μάλλον που έλεγε πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Αφρική το θέμα αυτό και ένας τρόπος να αποφύγουμε την ε, αύξηση της μετανάστευσης είναι να βρούμε, ε, να ενισχύσουμε την απασχόληση σε συγκεκριμένες χώρες. Και μάλιστα αναφέρθηκε ως παράδειγμα η Σενεγάλη. Και μάλιστα ε, με απασχόληση σε γεωργική εκμετάλλευση μπανάνας και προτάθηκε ως λύση για να περιοριστεί το πρόβλημα της μετανάστευσης. Τι γίνεται όμως με τη βιοπικιλότητα. Καταρχήν, ε, θέλουμε να έχουμε ασφαλή μετακίνηση του γενετικού υλικού, του βλαστοπλάσματος μπανάνας. Στη Λουβέν έχουμε 1060 ε, εισαγωγές, ε, καταχωρήσεις. Πολλές είναι in vitro, σωλήνες δηλαδή δοκιμαστικούς και επίσης έχουμε και κρυοσυντήρηση σε υγρό άζωτο, 1060 είναι τέτοιες εισαγωγές ε, πολλοί μίλησαν για το Σφάλμπαρτ, για την σημαντική προστατευμένη εκεί περιοχή. Ε, βέβαια δεν υπάρχει μηχανισμός προστασίας ε, σε σχέση με τέτοιες καλλιέργειες και εδώ μιλούμε για τη μπανάνα που έχουμε σημαντικό τμήμα του γενετικού υλικού της που διαφυλάσσεται σε κρυοσυντήρηση σε ε, ε, υγρό άζωτο. Επίσης έχουμε ηλιοφιλειωμένα δείγματα ε, φύλων για αναλύσεις ε, γονιδιακού υλικού DNA. Και επίσης έχουμε και μια ε, διαδικτυακή βάση δεδομένων, στην οποία δίνουμε στοιχεία και για το γενετικό υλικό. Ως συντονιστής ε, του Μούσα, της Μπανανιά, δηλαδή της οικογένειας αυτής, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει για την ομάδα μας αυτή, την κοινότητα των γενετικών πόρων, Χωρίς αυτή τη συνεργασία θα μπορούσαμε να συλλάβουμε όλη αυτή τη βιοπικιλότητα. Και τα γαλάζια, οι γαλάζιες που βλέπετε είναι τα εθνικά προγράμματα με τις συλλογέ τέτοιου γονιδιακού υλικού ή κάποιες ερευνητικέ προσπάθειες που γίνονται για τις γενετικούς πόρους της μπανάνας. Και μάλιστα στην Τσεχία, στην Ευρώπη, έχουμε το γονιδίωμα του, της μπανανιάς, και αυτό γίνεται σε επίπεδο ταξινομικής κατηγορίας, αποτύπωση του γονιδιώματος και με τη λέγη και το ζαμπλού προσπαθούμε να καθαρίσουμε το γενετικό υλικό, ώστε το υλικό που δίνουμε να είναι απαλλαγμένο από νόσους. Και μάλιστα φέτος είχαμε και μία σύμβαση με το Βοτανικό Κήπο κοντά στις Βρυξέλλες, ώστε να κρατούμε εκεί όλες τις ντόπιες ηθαγενείς ε, τύπους μπανάνας με τη μορφή σπόρων. Και ιδέα είναι να τις διανέμουμε στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες. Έχουμε ανάπτυξη παγκόσμιας τράπεζας σπόρων προκειμένου μετά τη, διατήρησή τους ε, να μπορούμε να αναπαράγουμε τους σπόρους. Βέβαια εκεί θα πρέπει να ενδύνουμε την έρευνα και σε ό,τι αφορά τη, τους σπόρους που διανέμουμε ε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία ώστε να εξυπηρετούμε το στόχο της βιοπικιλότητας. Πριν αναλάβω το συντονισμό για το Μουσανέτ, ήμουν σε έναν ε, παγκόσμιο όμιλο για την ε, γονιδιακή ακολουθία του, του γενετικού υλικού της μπανάνας. Και το κέντρο ε, προέλευση της μπανάνας είναι η Νοτιοανατολική Ασία, για όσους δεν το γνωρίσουν. Και τα βασικά είδη είναι το μούσα μπαλμπισιάνα και μούσα ακουμινάτα όλες οι μπανάνες που τρώμε έχουν κάποια διασύνδεση με αυτά τα δύο πρωτογενή ε, είδη ε, ποικιλία μπανάνας, μπαλμπισιάνα και νάτα. Έχουμε λοιπόν από την άποψη ανέβρεση της ακολουθίας του DNA, έχουμε κάνει ένα σημαντικό άλμα, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τα υποδέστερα είδη, το πανγονιδίωμα που λέμε δηλαδή, ε, να εξετάσουμε και τα γονίδια που μας ενδιαφέρουν και τα γονίδια που είναι στην πηγή της ε, μπανάνας που έχουμε σήμερα. Και αυτό κάνουμε στο Μομπελί, στην Νότια Γαλλία. Έχουμε αναπτύξει μία βάση δεδομένων που την αποκαλούμε η πύλη του πανγονιδιώματος. Η πρώτη εφαρμογή τέτοιων ε, δεδομένων γονιδιακής ακολουθίας ήταν δύο σημαντικές εφαρμογές. μάλιστα είχαμε το υλικό μας in vitro και η συλλογή του Λέβεν ε, υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Αλλά συστηματικά τροφοδοτούμε τη συλλογή αυτή με υλικό, αλλά χάρη στις πληροφορίες που έχουμε για την ακολουθία του DNA, έχουμε καταφέρει να διακρίνουμε μεταξύ του off-type, το κάτω ε, φυτό που είναι ε, το ίδιο, το ίδιο με το πάνω, το φυσιολογικό φυτό, με κάποιες όμως χρωμοσωμικές ανομαλίες. Και αυτό το βρίσκουμε με την καλλιέργεια του υλικού. Έτσι βλέπουμε ποιες είναι οι σωματοκλονικές παραλλαγές. Επίσης έχουμε εντοπισμό των γονιδίων χάρη στην τεχνική αυτή. Ξεκινήσαμε με, ένα με μια πιλωτική μελέτη για να κάνουμε διάκριση μεταξύ των μπανανών των, με σπόρο και των άσπορων. Φανταστείτε όταν χρησιμοποιείτε τέτοιο υλικό για μπανάνα, ξεκινάτε με την μπανάνα που έχει σπόρους και καταλήγουμε σε μια μπανάνα άσπορη που είναι το τελικό προϊόν. Οπότε είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη αυτή την, αυτόν τον εντοπισμό των γονιδίων που πρόσφατα δημοσιεύσαμε. Επίσης, προσαρμόζουμε τεχνική και σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ξηρασία, σε συνεργασία με την Λουβέν. Επίσης, ασχολούμαστε με σημαντικές νόσους και θα οργανώσουμε και ένα σεμινάριο στο Μαμπελιέ την επόμενη εβδομάδα για τι τεχνικέ μα αυτέ. Και εν να πω ότι η in situ διατήρηση λόγω ε, του, των περιορισμών της εξήτου διατήρησης είναι σημαντική. Καταρχήν έχουμε σωματοκλονικές παραλλαγές, όπως σας είπα, μεγάλες. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ε, το υλικό αναπτύσσεται στη φύση και μόνο μια επιτόπια διατήρηση θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα τώρα συνεργαζόμαστε με ένα κέντρο βιοπικιλότητας και βλέπετε τις αιστείες που είναι ε, σε κόκκινους κύκλους ε, στο χάρτη και προσπαθούμε με αυτή τη χαρτογράφηση των αισθειών, των βελτίωτων ποικιλιών, να δούμε όχι μόνο σε επίπεδο άγριων συγγενών, αλλά και σε επίπεδο ε, ντόπιων, αβελτίωτων ποικιλιών. Έχουμε την πρώτη μπανάνα, την πιο ε, ε, γνωστή και μία άλλη που είναι 100, 100 ε, φορές πιο θρεπτική από άποψη βιταμινών και μάλιστα είχαμε μια διανομή τέτοιων σπόρων στην Αφρική και με πολύ χαρά διαπιστώσαμε ότι στο Καμερούν σε ένα σεμινάριο που οργάνωσα ζήτησα από ένα μέλος, από ένα συμμετέχοντα στην οποία συμμετείχαν πολύ από τη Δυτική Αφρική και μάλιστα έχουμε μία από τις δέκα σημαντικότερες ποικιλίε στην αγορά. Ακόμη και χωρίς βελτίωση, δηλαδή μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ το γενετικό υλικό. Ε, αρκεί να είναι γνωστό το υλικό που υπάρχει παγκοσμίω. Τώρα έρχομαι και πάλι στο θέμα της αγροβιοπικιλότητας. Ελπίζω να σας έπεισε για το πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση της αγροβιοπικιλότητας και στην Διεθνή Αυτή Οργάνωση που, στην οποία συμμετέχω, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εταίρους για να αναπτύξουμε έναν δίκτυ αγροβιοπικιλότητας και να καταμετρούμε την αγροβιοπικιλότητα σε όλο το τροφικό σύστημα από τη γενετικούς πόρους παραγωγή, αγοράς και την κατανάλωση εντοπίζοντας ε, δηλαδή κινδύνους που σχετίζονται με χαμηλή ή φθήνουσα αγροβιοπικιλότητα και στον εντοπισμό ε, ευκαιριών για την αύξηση ή την ενίσχυση της αγροβιοπικιλότητας. Ο δείκτης αυτός ε, αγροβιοπικιλότητας στόχο έχει να μετατρέψει το σύστημα τροφίμων μας προωθώντας πιο συστήματα μεγαλύτερης βιοπικιλότητας σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, αγοράς, κατανάλωσης και για να διαφυλάξουμε την αγροβιοπικιλότητα θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και να επιτρέψουμε στον κόσμο να επωφεληθεί από αυτό το πλούτο και σήμερα και στο μέλλον. Συνεργαζόμαστε με πολλές κυβερνήσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης, αλλά και με ερευνητέ και επιχειρήσεις και πάλι εντός και εκτός της Ευρώπης για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Και τέσσερα μηνύματα θα ήθελα να σας, αναφέρω. Καταρχήν, η παραγωγή μπανάνας διατρέχει κίνδυνο λόγω της διάβρωσης της αγροβιοπικιλότητας σε όλα τα επίπεδα, από τη γενετική βιοπικιλότητα μέχρι τα τροφικά συστήματα. Δεύτερον, για να διαφυλάξουμε την αγροβιοπικιλότητα θα πρέπει να την καταμετρήσουμε, να τη διαχειριστούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε. Και πάλι ε, ο ρόλος εδώ των κοινοτήτων των γενετικών πόρων είναι πολύ σημαντικός. Και φυσικά θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σφαιρική ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω παγκοσμίων ε, τροφικών συστημάτων. Και τέλος, ε, η, η ομάδα μου, η οργάνωσή μου, η Bioversity International, ασχολείται με τα θέματα αυτά, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο αγροβιοπικιλότητας και για την επιστηστική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρου, Dr. Ρου. Πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Ε, εν ώψη των συζητήσεων λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η κυρία Μαγκίνες, η πρώτη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους α, τρεις α, ομιλητές μας. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, κάτι εντυπωσιαστεί με την εργασία που κάνετε και συνειδητοποιώ πόσο ζωτική σημασία είναι. Όπως είπε η κυρία Μπάρτ, θα πρέπει να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες. Το ερώτημά μου έχει να κάνει σε σχέση με τα ζητήματα in situ διατήρησης. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα προκειμένου να εντοπίσουμε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης ως περιοχές που θα μπορούσαν ε, να να προωθεί περισσότερο in situ διατήρηση των άγριων συγγενικών φυτικών ειδών. Κάθε φορά που προχωρούμε σε μια διαδικασία που εντοπίζουμε συγκεκριμένε περιοχές, αντιδρούν, για παράδειγμα, οι γεωργοί, οι αγρότες φοβούνται τις σχετικέ συνέπειε. Μήπως θα έπρεπε όμως εδώ πέρα να εκμεταλλευτούμε τις οικονομικές ευκαιρίες που μπορούν να δοθούν σε όσους κατέχουν τέτοια εδάφη σε περιοχές όπου θα μπορούσαμε να διασώσουμε αυτά τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Να τους δώσουμε δηλαδή ένα οικονομικό όφελος αν θέλετε. Αν δεν το πράξουμε αυτό, αν δεν καταφέρουμε να διατηρήσουμε ό,τι έχουμε εν situ, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Μπορούμε να να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα είδη στο εργαστήριο ή πρέπει να περάσουμε αναγκαστικά ούτως ή άλλως από ενσύτου του διατήρηση. Σας το συγγνώμη. Περιμένω από εσά απαντήσεις λοιπόν στα ερωτήματα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει πρώτος το λόγο. Νομίζω ότι όλοι μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό. συνήθως συγκεντρώνουμε τις ερωτήσεις από μερικούς ομιλητές, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε αμέσως, κανένα πρόβλημα. Μπορούμε αυτό να κάνουμε τώρα. Παρακαλώ. I think, uh... Κύριε Μπάρτ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι αγρότες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διαχείριση μεγάλων ε, αριθμών ποικιλιών και ειδών. Αν για κάθε είδος χρειάζεται να έχουμε εξίτου ένα ικανό δείγμα για τη διατήρηση, αλλά αυτό ε, ουσιαστικά είναι ανέφικτο, γιατί χρειάζεται κάθε χρόνο να ε, ανανεώνεται το υλικό, να ελέγχεται η ποιότητα, να διατηρούνται οι συλλογές και τα δύο χρειαζόμαστε. Για την in situ, την επιτόπια διατήρηση, ε, όντως χρειάζεται η συμμετοχή των αγροτών ή των γεωργών με κάποια αμοιβή όμως και μια προοπτική πιο μακροπρόθεσμη. από ό,τι ισχύει σήμερα. Όσον αφορά την in situ διατήρηση, προφανώς τη χρειαζόμαστε. Η ιδιαιτερότητα με την in situ δεν είναι ότι χρειάζεται αναγκαστικά να έχετε ένα μεμονωμένο είδος κάθε φορά. Έχουμε μια κοινότητα, αν θέλετε, ειδών που διατηρούμε εκ παραλλήλου. Αυτή είναι η προσέγγιση στην in situ διατήρηση. Και ο πιο εύκολος τρόπος να γίνει αυτό είναι στο πλαίσιο των ήδη καθορισμένων προστατευμένων περιοχών. Ήδη υπάρχει λοιπόν εκεί ένα δίκτυο προστευόμενων περιοχών. Μπορούμε απλώς να προσαρμόσουμε λίγο το σύστημα διαχείρισης που έχουμε, προκειμένου να καταφέρνουμε να καλύπτουμε και τα ίδια αυτά. Και θα έλεγα ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι τόσο δαπανηρή και μπορεί να γίνει. Στον Εμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχουμε μια τέτοια προστατευμένη περιοχή που την έχουμε εμπλουτίσει και με την πτυχή αυτή τη προστασία των άγρων συγγενικών φυτικών ειδών. Η εμπλοκή τώρα των γεωργών των αγροτών σαφώ είναι πολύ σημαντική. Αν δείτε για παράδειγμα τα 40 τέτοια είδη προτεραιότητας, τα περισσότερα από αυτά τελικά βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν είναι προστατευμένες. Τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη συνήθως τα βρίσκουμε σε περιοχές που βρίσκονται γύρω-γύρω από παραδοσιακές αγροτικές περιοχές. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους γεωργούς. Αυτό αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το μέλλον. Δεν χρειάζεται κανείς κατά αυτόν τον τρόπο να πληρώσει για την υποδομή μιας προστατευμένης περιοχής, αλλά θα πρέπει να δώσει ένα κάποιο οικονομικό αντίτιμο στους γεωργούς προκειμένου να προσαρμόσουν τις πρακτικές καλλιέργειάς τους γιατί να μην περιοριστούμε μόνο στην εξή του διατήρηση. Με αυτό που συμβαίνει με την εξή του διατήρηση είναι ότι χρησιμοποιείται ένα πολύ μικρό δείγμα και το βάζετε στην γονιδιακή τράπεζα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό της γενετική βιοπικιλότητα. Όταν μπαίνει επίση στη γονιδιακή τράπεζα, το δείγμα αυτό ψύχεται. Δεν έχει λοιπόν τη δυνατότητα να προσαρμόζεται φυσιολογικά και αυτόματα όπω θα έκανε αν ήταν ελεύθερο στη φύση. Θέλουμε λοιπόν όχι μόνο να έχουμε την in situ, επειδή μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τελικά ένα μεγαλύτερο δείγμα, αλλά επειδή το δείγμα αυτό μπορεί να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί πολύ καλύτερα και με πιο φυσιολογικό τρόπο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια στο εργαστήριο. Τώρα, σε σχέση με τα είδη τα οποία είδαμε, κάποια πρωτογενή είδη, όπως ε, στην περίπτωση της μπανάνας, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα αν ε, περιοριστούμε μόνο στην εξή του διατήρηση. Σε καμία περίπτωση να επιλέγουμε ανάμεσα στα δύο, θα πρέπει να συνδυάσουμε την εξή του και την in situ διατήρηση. Ευχαριστώ πολύ για το όσα είπατε, είπε κύριος Βάιτς, και για τη δουλειά σας. Δύο ερωτήσεις έχω. Μία ε, στον δόκτωρα Μάξτετ στην αρχή είπατε ότι υπολογίζεται, ε, θεωρείτε ότι ετησίως χάνουμε με την κλιματική αλλαγή 2% των ε, γεωργικών εκτάσεων. Έχετε συνυπολογίσει εκεί ε, τη διάβρωση, την καταστροφή του εδάφους ή την αλλά αύξηση της περιοδικότητας άλατος στα εδάφη. Ε, Μίλησατε για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το δεύτερο πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής, κυρία Μπάρτ, εσείς τώρα, για την προστασία της γεωργίας, ε, για ε, κάτι που γίνεται στη Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία και Ιταλία ήδη. Θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό και στον πρόεδρο και να το διαβιβάσω. Θα μπορούσαμε εδώ στην επόμενη ΚΑΠ να το φέρουμε στο επίκεντρο της προσοχής. Και μια ερώτηση προς τη δόκτωρα Μπάρτ. Ε, είπατε ότι χάσαμε 70% ε, του πληθυσμού των εντόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει καμία σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέιτς. Παρακαλώ κύριε Μπάρτ ή όποιος θέλει. Θα απαντήσω εγώ στην πρώτη ερώτηση. Το 2% δεν περιλαμβάνεται άλλα είδη διάβρωσης. Αυτό προστίθεται στην κανονική διάβρωση το 2% και δεν είναι από το κεφάλι μου τα στοιχεία, αλλά από το Διεθνές Πάνελ Κλιματικής Αλλαγής. Στην τελευταία έκθεση αυτό το ποσοστό προέκυψε. Νομίζω. Ε, γίνεται μεγάλη συζήτηση. Ε, πού οφείλεται ε, ε, το, η απώλεια και η εξαφάνιση των εντόμων που κάνουν την επικονίαση. Πολλοί είναι οι παράγοντες, κλιματική αλλαγή, ε, γεωργικές πρακτικές, μεταξύ άλλων. Αλλά τελικά αυτό είναι απειλή και για την αποτελεσματική διατήρηση in situ. Γιατί χρειαζόμαστε τα ε, έντομα της επικονίασης, ιδιαίτερα για τα ψυχανθή, και άλλα είδη. Αν υπάρχει μια περιοχή λοιπόν που θα χαρακτηριστεί ε, περιοχή στρατηγική για διατήρηση in situ, μήπως να βάλουμε και τίποτα έντομα εκεί για να κάνουν την επικονίαση. Δεν θα ήταν παράλογο. Για να έχουμε καλύτερες στρατηγικές διατήρησης των ειδών. Η κυρία Μακιντάρ. Ε, Σας ευχαριστώ. Και θερμότατα ευχαριστώ προς τους καλεσμένους εμπειρογνωμονές μας. Όταν προδάκουσα για την πρόταση αυτή τη δημόσια εκρόση, σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Ήταν συναρπαστική η ακρόαση αυτή και πραγματικά ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για μας να φτάσουμε σε τόσο ευρυθείς γνώσεις και θα μας βοηθήσουν και στο μέλλον. Πριν από ένα χρόνο και είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλία στην Επιτροπή, για την οποία ήμουν εγώ εισηγήτρια, για τις τεχνολογικές λύσεις για το μέλλον της γεωργίας. Και αφιερώναμε ένα ολόκληρο τμήμα της έκθεσης στην γενετική βιοπικιλότητα. Είναι ένας τομέας που δεν συγκεντρώνει τη δέουσα προσοχή. Εσείς όμως μας επισημάνατε τον άμεσο σύνδεσμο της επιστηστικής ασφάλειας και της γενετικής ποικιλομορφία. Ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πια λοιπόν αυτή τη γενετική ποικιλομορφία γιατί είναι άρρηκτα δεμένη, συνδεδεμένη με την επιστηστική ασφάλεια. Δυστυχώς η κυρία Μαγκίνης χρειάστηκε να φύγει, αλλά ε, εγώ θα ήθελα να επεκτείνω λίγο τα δικά της ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την ιδέα της ε, διατήρησης επιτόπου in situ, τα διάφορα συστήματα που έχουμε στην ΚΑΠ και τα κίνητρα που δίνονται για αγροπεριβαλλοντικά έργα, ίσως θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε ώστε να επιτρέψουμε διατήρηση in situ τέτοιων άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ε, φυτών και ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών που θέλουμε να διαφυλάξουμε. Αυτό είναι μια πιθανότητα για να δώσουμε κίνητρα στους αγρότες ότι αξίζει πραγματικά να ασχοληθούν και με αυτό, με την διατήρηση in situ. Γενικώ θέλουμε ερευνητικά κονδύλια να αφιερώνονται σε τεχνολογικές βελτιώσεις και γενικώ στην γεωργία και την καλλιέργεια παρακευευτικών, αλλά όπως είπατε υπάρχουν πολλά κενά σε αυτή τη χρηματοδότηση. Εσείς ως εμπειρογνώμονες, τι θα θέλατε να χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα, δηλαδή ποιο κενό να γεφυρώσουμε κατά προτεραιότητα στο χρηματοδοτικό κενό που έχουμε στην έρευνα. Παρακαλώ. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα που θα πρέπει να αφιερώνει η Γεωργία στην διατήρηση in situ. Όντως, συμφωνώ και μάλιστα έκανα λόμπι στη Natural England που καταβάλει αυτές τις πληρωμές τους αγρότες να συμπεριλάβουν και άγρια συγγενή και μάλιστα η διατήρηση in situ είναι ένα από τα κριτήρια που δημιουργούν την επιλεξιμότητα για τη χρηματοδότηση στην κυβερνητική. Και ακριβώς αυτό εννοούσα όταν είπα ότι τα περισσότερα άγρια συγγενή βρίσκονται εκτός προστατευμένων περιοχών, γύρω από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οπότε η καλύτερη ε, ιδανική τοποθεσία είναι εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για επιτόπια διατήρηση. Τώρα για τα, τα κενά, τα χρηματοδοτικά κενά στην έρευνα. Ναι, τι να πρωτοκαλύψουμε στην έρευνα. Στη δικιά μου περίπτωση και στην ομάδα, την συνεταιριστική ομάδα για, την, για τις φυτικούς γενετικούς πόρους. Έχουμε πολλές επιδοτήσεις ε, και έχουμε αντιληφθεί τι χρειάζεται σε διατήρηση in Ξέρουμε πού θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειες. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε στη δράση. Και αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, θα πρέπει κυρίως ε, να αφιερωθούν στη δημιουργία κάποιων ε, δομών διακυβέρνησης, διαχείρισης, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν οργανώσεις όπως η Natura 2000 που έχουν τέτοιες ε, δομές διακυβέρνησης. Οπότε αν έχουμε ένα δίκτυο τέτοιων ε, in situ τοποθεσιών διαφύλαξη τέτοιων ειδών θα πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη. Δεν ξέρω, το ECPGR ε, δεν ξέρω αν μπορεί να αναλάβει αυτό το, το, το ρόλο γιατί δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για να προσφέρει αυτές τις δομές διακυβέρνησης και να ε, μπορέσει να συντονίσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διατήρηση in situ των άγριων συγγενών. Η κυρία Αγγιλέρα, έχουμε τόσους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω ένας ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Το θέμα αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς και γι' αυτό πολλές φορές παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη ε, όλα αυτά τα στοιχεία γιατί δεν τα γνωρίζουμε για τη βιοπικιλότητα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Να αρχίσω από αυτό το τελευταίο που είπατε. Και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Για να μπορεί κάποιος να κάνει αυτή τη διατήρηση, τι χρειάζεται. Πρέπει να διατηρηθούν φυσικά κάποια ε, είδη, αλλά in situ, για την επιτόπια διατήρηση δεν θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στα πλαίσια του δικτύου Natura 2000, στους εθνικούς δρυμούς, τα ε, φυσικά πάρκα που είναι προστατευόμενες περιοχές και ζώνες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ήδη με κονδύλια που προβλέπονται από το δίκτυο Natura 2000. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο εντός αυτών των χώρων Εκτός της υγιεινής γεωργικής πολιτικής, στο περιβάλλον τώρα, στο Natura 2000, δεν υπάρχει δυνατότητα ε, σε αυτές τις προστατευμένες περιοχές να υπάρξει κάποια ειδική μέρημνα γι' αυτό. Το σκέφτηκα μετά από αυτά που μας είπατε, γιατί κατανοώ ότι πρέπει να γίνει και είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Εγώ δεν βλέπω τεράστια προθυμία από τους αγρότες ο αγρότης επάγγελμα κάνει για κέρδος. Ακόμα και αν χρειάζεται βιοπικιλότητα για το μέλλον, δηλαδή ότι θα πρέπει ο κάθε γεωργός να φροντίζει, να βάζει το λιθαράκι του στη βιοπικιλότητα, θα πρέπει να έχει και κάποιο κίνητρο για να τον βοηθήσουμε, να τον παροτρύνουμε να το κάνει. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να βρούμε κονδύλια από τα εθνικά πάρκα στην Ισπανία και μόνο. Είναι πολύ αναπτυγμένο αυτό το δίκτυο. Ενδεχομένως να βρούμε τα λεφτά από εκεί. Θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό. Άλλη ερώτηση, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο ενδεδειγμένος να απαντήσει. Αναφερθήκατε ε, στο εξής, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να αναμίξουμε ε, τα άγρια είδη με τις συμβατικές ποικιλίε τις ήμερες, με διασταύρωση. Αυτή η διασταύρωση των ειδών είναι γενετική τροποποίηση ή άλλο πράγμα. Δεν τα ξέρω, απόλυτη άγνοια δηλώνω. Ε, το ξέρω ότι τρομάζει ε, ο όρος γενετικά τροποποιημένος, όχι εμένα, τρομάζει γενικά τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η τεχνική διασταύρωση των ειδών. Ενδιαφέρον θα ήτανε για να δούμε πώς μπορούμε να διασταυρώσουμε άγρια με ήμερα ήδη. Ε, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο σας ερώτημα. Όπως σας είπα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε για την εργασία στα πλαίσια του δικτύου Natura 2000 είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί ήδη στα πλαίσια συγκεκριμένων κοινοτήτων ειδών όπου δεν περιλαμβάνονται τα άγρια συγγενικά φυτικά είδη. Πάντως, αν καταφέρναμε πραγματικά όσοι διαχειρίζονται τα πάρκα Natura 2000 να εντάξουν σε και σε αυτά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν με τα άγρια γενικά είδη, τότε τα πράγματα ήταν καλύτερα. Αλλά ακόμα και αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Στο Μένο Βασίλειο, όταν άρχισα να πρωτομιλώ σε διαχειριστές τέτοιων εθνικών πάρκων στο Μένο Βασίλειο για τα άγρα γενικά είδη, κατευθείαν είπαν ότι δεν ενδιαφέρονται. Δεν μας ενδιαφέρουν, είπαν οι καλλιέργειες. Επίσης, με τους περισσότερους χώρους Natura 2000, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην απουσία ή την παρουσία κάποιων ειδών. Με αποτέλεσμα τελικά να μην υπάρχει μία πλήρη κάλυψη της βιοπικιλότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι θεωρητικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο Natura 2000. Είναι σίγουρα καλή ιδέα, αλλά όχι μόνη καλή ιδέα που θα μπορούσαμε να είχαμε. για το πρώτο σας ερώτημα όσον αφορά την διατήρηση σε εθνικά πάρκα προστατευμένα. Στην Παππούα Νέα Γουινέα, ε, μία από τις εστίες διατήρησης είναι εθνικό προστατευόμενο πάρκο, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όντως την επιλογή αυτή και θα έλεγα και κάτι ακόμα. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με βοτανικούς κήπους οι οποίοι ε, βρίσκονται κοντά στα πάρκα αυτά και εκεί πέρα θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε περισσότερο σπόρους. όσον αφορά την γεωργία. Στα πλαίσια του, του δίκτυα αγροβιοπικιλότητας, ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους γεωργούς στα συστήματα τα επισητιστικά. Η Ρόζαλιν Ρέιμαντς, μία συνάδελφός μου, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά και θα ήταν η πλέον αρμόδια για να σας δώσει πιο συγκεκριμένε ε, ε, πληροφορίες. Εκεί πέρα ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδυάσουμε γεωργικές δραστηριότητες και διατήρηση άγρων συγγενικών ειδών. Όσον αφορά τη διασταύρωση ειδών, συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα μπορούσε τελικά να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν προχωρούμε κυρίως στην ενσύ του διατήρηση δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια διασταύρωση. Καμία περίπτωση πάντως το φυτό το οποίο προκύπτει δεν θεωρείται γενετικά τροποποιημένο φυτό. Δεν ξέρω αν η συνάδελφος θέλει να πάρει το λόγο. Thank Ευχαριστώ. Όντως, από τη μία είναι σημαντικό να καταμετρούμε και να παρακολουθούμε ε, αυτό το γρασιγενή και να δίνουμε κίνητρα σε όλο το σύστημα το τροφικό για τη διατήρησή του και συνεργαζόμαστε και με τον ιδιωτικό κλάδο για το θέμα αυτό. Και με το χρηματοπιστωτικό κλάδο, με τους επενδυτές, για να δημιουργήσουμε και οικονομικά κίνητρα στο σύστημα τροφίμων για ενίσχυση της βιοπικιλότητας των συστημάτων μας. Ε, υπάρχει το θέμα της ε, διαχείρισης γενετικών πόρων, της βιοπικιλότητας, αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, παραγωγής και των αγορών. Θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να δράσουμε ταυτόχρονα και επίσης να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές. Γιατί αν ε, γίνει πιο συνειδητοποιημένος από αυτήν την άποψη ο καταναλωτής, θα γενικευτεί αυτή η λύση. Και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε και τέτοιου είδους κίνητρα, δρώντας σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να, να πω κάτι για τα δύο τελευταία σχόλια. Καταρχήν, η αποτελεσματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ΣΥΤΟΥ θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη στα μελλοντικά μας προγράμματα για να ξέρουμε πόσα από αυτά θα κρατήσουμε και στο μέλλον. Επίσης, πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε και την περιφερειακή εφαρμογή, όχι μόνο την πανευρωπαϊκή. Γιατί πολύ συχνά η ίνση του διατήρηση ε, γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Ε, μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Το περιφερειακό σκέλος είναι πολύ σημαντικό. Για το πώς λειτουργεί αυτή η διασταύρωση και αν θεωρείται απαλλαγμένη από γενετικό τροποποιημένο οργανισμούς. Ναι, είναι απαλλαγμένο, δεν είναι γενετική τροποποίηση αυτή. Και ιδιαίτερα αν μιλούμε για ανθεκτικότητα σε νόσους ή ποιότητα, μπορούν κάποια γνωρίσματα από άγρια συγγενή να συμπεριληφθούν σε, στα ήμερα είδη, στις ήμερες ποικιλίε. Αλλά είναι μακρύς ο δρόμος ε, τέτοιου είδους διασταύρωση. Αν τα καταφέρουμε βέβαια θα είναι πολλά τα θετικά και το ωφέλη. Ο κύριος Αντριέ είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτή και τους τρεις ομιλητές για την ποιότητα των παρουσιάσεων και την ακρίβεια του περιεχομένου. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή ε, που προετοιμάζουμε τη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το μόνο ίσως κάπως ε, δυσάρεστο ε, είναι η μικρή παρουσία των Ευρωβουλευτών, ε, γιατί θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Και μας φέρετε αντιμέτωπους με τις ευθύνες μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς είμαστε πολιτικοί ε, που βάζουμε το λιθαράκι μας ε, στην ε, αλλαγή της νομοθεσίας για να καθορίσουμε κάπως ε, τα πράγματα του κόσμου που μας περιβάλλει. Και εδώ πρόκειται για κοινή κληρονομιά που δεν είναι ίσον σημασία η βιοπικιλότητα. Και τη στιγμή που καλούμαστε να νομοθετήσουμε επηρεάζουμε αυτή τη βιοπικιλότητα γιατί είμαστε και η Επιτροπή Γεωργίας. Και ε, πραγματικά είναι συγκεκριμένη αυτή η αναφορά σας. Μας παραπέμπεται στον πλούτο ε, ε, αυτών των ποικιλιών που αγνοούμε εμείς. Και τελικά τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η γεωργία στο περιβάλλον. με την πάροδο των ετών δεν είναι καθόλου ουδέτερη. Υπήρξε μια ολόκληρη εξέλιξη της γεωργίας ή των διαφόρων μορφών καλλιεργιών και του γεωργικού προτύπου ε, και σε καμία περίπτωση δεν ήταν ευκαταφρόνητος αυτός ο αντίκτυπος ε, στην επιδείνωση και τα καταστροφή τελικά του ε, περιβάλλοντος και του, του βιοτόπου. Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το μοντά της γεωργίας, γιατί δεν είναι ακόμα ένας κλάδος της οικονομίας. Επηρεάζει βεβαίως και την δημόσια υγεία, αλλά το περιβάλλον, τα εδάφη, τον αέρα, τον ατμοσφαιρικό, το νερό κτλ. Άρα, τι μοντέλο γεωργίας θα επιλέξουμε που έχουμε ήδη επιλέξει, που θα αλλάξουμε στο μέλλον, γιατί ε, είναι μια διάδραση αυτή και με ε, το φυσικό περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα. Και πώς αυτό εντάσσεται, ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε την υπερπαγκοσμιοποίηση και την υπερσυγκέντρωση των ε, καλλιεργειών και δεν λαμβανόταν αρκετά υπόψη το ε, περιβάλλον και ο περίγυρος. Μα αυτή είναι η γεωργία, έχει μια ομορφιά να δίνει τροφή ε, στον πληθυσμό της γης άνδρες και γυναίκες. Τα είπατε κι εσείς όλοι και η κυρία Μπάρτ το πιο εύκολο, ε, ακούσαμε για, για γενετικά τροποποιημένα τώρα, το πιο εύκολο μοντέλο στη γεωργία ήταν να χρησιμοποιούμε ε, γεωργικά εφόδια χωρίς να έχουμε υπόψη μας τη γεωπονία με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Θα πρέπει λοιπόν η γεωπονία να πονάει τη γη και να την, να την ε, καλλιεργεί για να μην καταστρέφουμε τη βιοπικιλότητα αλλά να υπηρετούμε το δημόσιο κοινό συμφέρον. Είπατε ότι οι χορτονομές και τα λιβάδια, οι λιμόνες που έχουν διάφορα ε, φυτά ε, είναι τα πιο παραγωγικά. Γιατί έχουμε εγκαταλείψει λοιπόν την αμύψη σπορά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Θέλουμε λιμόνες φυσικούς, θέλουμε εναλλαγή καλλιεργειών ακριβώς σε αμύψη σπορά. Ε, το είπατε πολύ για το περιβάλλον. Εδώ πήραμε μια απόφαση για τις ε, περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος επιφάνειες όπου απαγορεύονται τα ζυζανιοκτώνα. Χαμός έγινε. Ε, με πολύ μικρή διαφορά πέρασε και μικρή πλειοψηφία. Ε, καταλαβαίνουμε ποια είναι η συνειδητοποίηση αυτών των θεμάτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που καλούμαστε να αλλάξουμε προσανατολισμό, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το γεωργικό μας μοντέλο. Μπορούμε και ανταγωνιστικοί να είμαστε, σεβόμενοι το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Για να έχουμε λοιπόν ένα τρόπο παραδοσιακής καλλιέργειας, γεωπονίας, μια χρηστή διαχείριση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αυτή τη γεωργία και όπως εξελίχθηκε καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον. Και πολύ σωστά αναφέρεστε στα έντομα της επικονίασης που αν καταστραφούν και αφανιστούν αύριο θα καταστραφεί ολόκληρη και η γεωργία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλους ομιλητέ στον κατάλογο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο για τι τελικέ απαντήσει ε, στι ερωτήσει του κυρίου Αντριέ, για να ολοκληρώσουμε τη δημόσια μας ακρόαση. Ποιο από όλου θέλει να απαντήσει. Κυρία Πάρθ ή κάποιο άλλο. Okay. Uh, Νομίζω ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ξανά την ε, γεωργία να συμπεριλαμβάνει στοιχεία προστασίας ε, της γενετικής ποικιλομορφίας. Να μπορεί να χρησιμοποιεί η κλασική, αν θέλετε, γεωργία τα στοιχεία αυτά και να μπορεί επίσης να διασφαλίζει τη γενετική ποικιλομορφία για το μέλλον. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μια γενετική φυτική κληρονομιά, αλλά για νέα στοιχεία παραγωγής, τα οποία θα μας επιτρέψουν να διασφαλίσουμε την επισητιστική ασφάλεια που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Και ελπίζω ειλικρινά ότι θα καταφέρουμε να έχουμε στο μέλλον και πολιτικές οι οποίες θα είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον όσον αφορά τη γεωργία και, θα, και ελπίζω να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο και την θετική επίδραση των εντόμων. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Προφανώς το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο θα πρέπει να αναλάβουμε δράση όσον αφορά την γενετική ποικιλομορφία, γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για αγροβιοπικιλότητα, ποικιλότητα δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει προφανώς να μετασχηματίσουμε τον τρόπο που παράγουμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την διοπικιλότητα. Και προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε όσους θέλουν διατηρήσουν τη βιοπικιλότητα αυτή όχι μόνο σε επίπεδο συντήρησης και διατήρησης, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο. Εκεί θεωρώ ότι μπορεί να εμπλακεί περισσότερο η γεωπονία. Μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ασχολούνται με τη διατήρηση. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, να προωθήσουμε πιλωτικά προγράμματα, που θα θέλαμε στο μέλλον να μπορούν να εφαρμοστούν σε πιο ευρία βάση για μένα πραγματικά το μυστικό έγκυται στα κίνητρα τα οποία θα δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Διεκπερώσαμε το πρόγραμμά μας. Ε, νομίζω ότι όντως πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ήταν πολύ καλή αυτή η συζήτηση. Γιατί μας δίνει και τροφή για σκέψη κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Και ήταν πολύ σημαντικό το σχόλιο του κυρίου Αντρία. Βέβαια, εκείνο καλύτερα θα ήταν ορμόδιο να σχολιάσει περαιτέρω αυτά που είπε και να δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για τη σκέψη του ω προ το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική. Πραγματικά ήταν ε, συναρπαστικέ οι ομιλίε που ακούσαμε. Σα ευχαριστώ θερμά εξαιρετικές και πραγματικά ε, μας έδωσαν ε, πολλές χρήσιμες πληροφορίες και είναι πηγή έμπνευσης και για τις ε, περαιτέρω συζητήσεις μας για το μέλλον της ΚΑΠ. Η Επιτροπή μας είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα, τα θέματα της βιοπικιλότητας και πιστεύω ότι και η Γεωργή μας το ίδιο. Για να δούμε πώς τα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια που ετοιμάζονται τα κράτη-μέλη θα εντάξουμε και αυτή τη διάσταση. Επόμενη εβδομάδα ε, είναι εβδομάδα του Στρασβούργου. Δεν προβλέπεται συνεδρίαση πριν τις διακοπές, οπότε σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους, ε, το προσωπικό, τους διερμηνείς. Η επόμενη μας συνεδρία θα γίνει στις 11 Ιανουάριου. Α, θα συνεδριάσουν και οι συντονιστές στο Στρασβούργο όμως. Αυτά, σας εύχομαι καλή επάνωδο. Λυπάμαι που χρειάστηκε να σας κουβαλήσω εδώ πέμπτη απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο γιατί ήταν πολύ σημαντική ακρόση και να είστε βέβαιοι το περιεχόμενο θα το διαβάσουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Α, και καλωσορίζουμε και τον κύριο Τεγκάστρο ήταν πραγματικά θαυμάσιο αυτό το θέμα. Πολύ καλή και φαντάζομαι περισσότεροι είναι κάπως εξοικειωμένοι. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν οι εμπειρογνώμονες μας. Σας ευχαριστώ και χαίρετε. Καλό βράδυ.